για εγκλήματα που σχετίζονται με την Πανίδα και τη Χλωρίδα. Με τι? Ξονόματος ε, του συντάκτη ο κύριος Γκερμπράντι για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από δύο χρόνια εγώ είχα ανησυχήσει από κάτι νούμερα για τεράστια αύξηση εμπορίου ε, των κεράτων των ρινόκερων στην Νότια Αφρική και φαίνεται πως αυξάνονται τα νούμερα και από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο το η μύτη του ρινόκερου αλλά και 30-40 ελέφαντες ε, που σκοτώνται κάθε χρόνο για το ελεφαντόδοντο και αλλά και τίγρης, ε, ερπετά, αρπακτικά, ακόμα και δέντρα η φύση από ό,τι φαίνεται πλέον ε, αποτελεί αντικείμενο τραγικής εκμετάλλευσης ε, και ειδικά αυτό στην Νοτιοανατολική Ασία όπου υπάρχουν παράνομα προϊόντα από την φύση αξίας πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μιλάμε για το τέταρτο παράνομο εμπόριο μετά τα ναρκωτικά, τις απομιμήσεις και το εμπόριο ανθρώπων έχουμε το εμπόριο αυτό που σας ανέφερα. Και καταρτήσαμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης το οποίο υποβάλαμε και χαίρομαι για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτησε κάποια στοιχεία του μεταξύ άλλων. Ε, καταλήξαμε σε μια συμφωνία με την Κίνα για συνεργασία για την καταπολέμηση του εγκλήματος αυτού. Αλλά κύριε Πρόεδρε βεβαίω δεν επαρκούν καθόλου αυτά τα μέτρα και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία του 2013. Και πέρσι δυστυχώς το έγκλημα αυτό αυξήθηκε εκρηκτικά. Πάνω από 100 μύτες ε, ρινό καιρού το 2009, 300 πέρσι ε, και πάμε από ό,τι φαίνεται για ένα νούμερο που θα προσεγγίζει τα χίλια. Πρέπει όλοι να βοηθήσουν. Νίκιο, δασοφύλακες, ε, Interpol, ε, το πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ και πάρα πολλοί άλλοι. Οπότε το συμπέρασμα είναι σαφές. Εάν δεν κινηθούμε γρήγορα με ε, δραστικά μέτρα για να σταματήσουν αυτές τις παράνομες πρακτικές, προσεχώς θα έχουν εξαφανιστεί τα πιο εμβληματικά είδη άγριας ζωής. Γι' αυτό αναλάβαμε την ε, πρωτοβουλία για αυτή την προφορική ερώτηση και ψήφισμα, επειδή είναι μεγάλος ο ρόλος της Ευρώπης. Το θέμα δεν είναι μόνο η Αφρική και η Ασία και θα σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια ηθική υποχρέωση για να σταματήσει αυτή η μαζική σφαγή. Και δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Και δεύτερον, ε, τα κράτη μας παίζουν ένα σημαντικό ρόλο ως προορισμός και ως ε, κέντρο διαμετακόμισης ε, στην ε, Ολλανδία. Πέρσι πιάσαμε ένα φορτίο τεράστιο με τέτοια είδη. 680 κιλά παράνομα κοράλια σε ένα πακέτο ή χιλιάδες ε, νεκροί απόκαμπη επίσης ε, αντικείμενο παράνομης εμπορίας. Οπότε υπάρχει αρκετά μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω την Κομισιόν για το ρόλο που παίζει. Κατόπιν, κύριε Πρόεδρε, το έγκλημα αυτό έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Αποσταθεροποιούνται ολόκληρες περιοχές. Ε, το χρήμα είναι μεγάλο κίνητρο. Και δισεκατομμύρια σε αναπτυξιακή βοήθεια πάνε χαμένα τι πρέπει να συμβεί. Πρώτα απ' όλα λοιπόν είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη-μέλη να καταλήξει σε ένα δικό της σχέδιο δράσης. Συγκεκριμένο και φιλόδοξο. Σε κράτη-μέλη επίσης. Και για να ανοιχνεύσουμε τις διαδρομές αυτές, αλλά βεβαίως και για να υπάρξει μεγαλύτερη δημιουργία από πλευράς ποινικού δικαίου. Πρέπει να το δούμε αυτό ως αυτό το οποίο είναι, δηλαδή οργανωμένο έγκλημα. και να αποδοθεί πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα σε αυτό. Επίση, πρέπει να δημιουργηθεί εντό τη Europol μια μονάδα εγκλήματος κατά της άγρια ζωή. Τόσο σημαντικά είναι τα πράγματα. Επίσης οι εμπορικέ συμφωνίε πρέπει να έχουν τέτοιε ρήτρε, Να υπάρχει δηλαδή μια αιρεσιμότητα που θα αφορά τη συνεισφορά στην καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος. Επίση, το ψήφισμα αναφέρεται κύριε Πρόεδρε πως η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη πρέπει να δημιουργήσουν ένα καταπίστευμα για να χρηματοδοτηθεί αυτή η προσπάθεια. Και ολοκληρώνω εδώ πέρα. Τι κάνουμε δηλαδή, τι νόημα έχει να λέμε ότι είμαστε πολιτικοί και να παρατηρούμε άπραγη το διαγούμισμα της φύσης πραγματικά για να κερδίζουν δισεκατομμύρια διάφοροι εγκληματίες. Τίποτα δεν αξίζουμε λοιπόν ως πολιτικοί εάν δεν κάνουμε τίποτα. Υποθέτω λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα συμφωνήσουν με το Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο δράσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε εξ ονόματος Κομισιόν. Καλωσορίζω τον κύριο Ποτότσνικ και έχετε τον λόγο. Mr. President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γερμπράντη και όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι ευγνώμων για αυτή την πρωτοβουλία να θέσετε το θέμα της ε, καταπολέμησης του εγκλήματος εις βάρος των αγρίων ε, ζώων. Δυστυχώς έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Πρόκειται μία, από για μία από τις πιο επικερδείς εγκληματικές δραστηριότητες παγκοσμίως και ε, καταστρέφει τη βιοπικιλότητα καθώς και την ύπαρξη εξαλείφει ε, πολλά βασικά είδη, άγρια είδη. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την προέλευση καθώς και τις χώρες διαμετακόμισης και τις χώρες προορισμού αυτών των ειδών. Εμείς και με την ΣΥΤΕΣ συνεργαζόμαστε ε, για αντιμετώπιση εμπορίου ειδών υπό εξαφάνιση. Έχουμε υποβάλει μία πρόταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνουμε πλήρες μέλος του ΣΥΤΕΣ και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να συνενέσει πριν από τις εκλογές. Επίσης, ανακύπτει το ζήτημα της αντιμετώπισης ε, της παράνομης εμπορίας των αγρίων ειδών. Δηλαδή αυτό το είδαμε τον Κινέζο ομόλογό μου, και επίσης θεωρούμε ότι οι ΣΥΙΤΕΣ και ε, αφρικανικές χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν επί του θέματος ε, γιατί είχαμε 12,3 ε, εκατομμύρια μέσα στα πλαίσια ενός project για να αντιμετωπίσουμε το έγκλημα κατά των ελεφάντων ιδιαίτερα. Να καταπολεμήσουμε την παράνομη θύρευση των ε, ελεφάντων και άλλων ειδών. Όμως, ε, δυστυχώς, ε, το εμπόριο αυτό είναι ιδιαίτερα αποδοτικό, δηλαδή... δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κέρας του ρινόκερου ε, είναι πιο επικερδές από την κοκαίνη. Είναι πολύ ε, εύκολο να γίνει λαθρεμπόριο και δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά μέτρα αναχέτησης. Δυστυχώς η εμπορία του ελεφαντοστού έχει αυξηθεί και ε, δυστυχώς και η Ευρώπη είναι ήπειρος διαμετακόμισης. Η διαφθορά βοηθά την λανθρεμπορία καθώς και το οργανωμένο έγκλημα το οποίο ε, διακυβεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα. Χρειαζόμαστε αναγνώριση της απειλής ε, αυτής της ε, παράνομης εμπορίας των αγρίων ειδών θα πρέπει να κινηθούμε σε, σε επίπεδο υπουργών, τελωνιακών αρχών, δικαιοσύνης, ΜΚΟ και ιδιωτικού τομέα. Όλοι έχουν να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ε, ρόλο. Το ερώτημά σας με αίτηση προφορικής απάντησης μπορεί να οδηγήσει σε απαντήσεις γιατί και οι ΙΠΑ θα δεσμευθούν κατά της ε, λαθρεμπορίας αγρίων ειδών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προβάλλει μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της λαθροθυρίας και τον επόμενο μήνα θα υποβάλουμε μία πρόταση μαζί με την Επίτροπο Μάλστρομ σε στενή συνεργασία και με άλλους επιτρόπους και με τον Επίτροπο Πίμπαλξ για να προβάλλει ένα νέο μέσον προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα επίγον ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε παγκοσμίω. Με βάση τα ήδη υπάρχοντα ευρωπαϊκά μέτρα θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και παγκοσμίω. Και επίσης θα δούμε πώς θα προσεγγίσουμε το θέμα μελλοντικά σε σχέση με την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των αγρίων ειδών. Ε, τα δεδομένα είναι διαφορετικά, γι' αυτό θα πρέπει να προβάλλουμε νέες ιδέες για να αντιμετωπίσουμε και θέματα ειρήνης και σταθερότητας και να προβάλλουμε άλλες πηγές βιωσιμότητας. Γι' αυτό θα θέλαμε οι εμπλεκόμενοι φορείς να μας ε, ανοίξουν νέες οδούς για πραγματική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα διοργανωθεί μια διάσκεψη στις 10 Απριλίου το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οδηγεί σε μια δημόσια συνειδητοποίηση του ζητήματος και η Επίτροπος Μάλστρομ και εγώ προσβλέπουμε με ανυπομονησία τη συζήτηση μαζί σας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση της λαθρεμπορίας και θύρευσης των αγρίων ειδών. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Περνάμε στους ομιλητές των ομάδων. Για τρία λεπτά τον λόγο έχει για το ΕΛΚ η κυρία Γιόρνταν. Ευχαριστώ. πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον εισηγητή και την Επιτροπή για το θέμα. Μιλάμε για ρινόκερους, ελέφαντες, τίγρεις, χελώνες, και ίσως ε, δεν το έχουμε αντιμετωπίσει επαρκώς το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό διότι αυτή η παράνομη εμπορία μπορεί να υπονομεύσει το κράτος δικαίου και την βιοπικιλότητα. Αυτές οι εγκληματικές δραστηριότητες προωθούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο σε τρίτες χώρες. Και αυτό το βλέπουμε από τις κατασχέσεις που γίνονται μέσα στα πλαίσια της Σύμβασης ΣΥΤΕΣ. Εγώ έχω εξετάσει τα στοιχεία του 2012 και είδα ότι είχαμε 799 αιτήσει κατασχέσεων. Τα περισσότερα προϊόντα ε, προορίζονταν για ιατρική χρήση. Υπάρχει και το θέμα του ελεφαντοστού. Η Ευρώπη μπορεί να είναι και τελικός ε, προορισμός ή χώρος διαμετακόμισης. Γι' αυτό θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό όμως που χρειαζόμαστε είναι μια κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη ως προς την ομοθεσία τους για να είναι συνεπής και ομοιογενής και να υπάρχει παρόμοιο επίπεδο ε, κυρώσεων. Έτσι ώστε να μην ε, ανοίγουμε την ε, οδό ώστε να γίνεται ε, λαθρεμπόριο σε ορισμένες χώρες. Γι' αυτό και η ομάδα μου δεν υποστηρίζει τη δημιουργία νέων ε, ταμείων ή μέσων για αυτό το στόχο. Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε διεθνώς τη διάσταση του ζητήματος. Η σύμβαση του ΣΥΤΕΣ ισχύει από το 1975 και πέρσι τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι το έγκλημα κατά των άγριων ειδών είναι εξίσου σοβαρό ε, όσο, και το έγκλημα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, με τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτό το τόνισε και ο πρόεδρος Ομπάμα. Θα πρέπει όμως να δράσουμε παγκοσμίως, να είμαστε δραστήριοι και να υποστηρίξουμε, όπως και η ομάδα μου, αυτό το ψήφισμα και πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε το έγκλημα αυτό, τη διάστασή του. Επίσης δεν υπάρχει εμπόριο χωρίς ζήτηση και γι' αυτό θα πρέπει να τονίσουμε την ε, συνειδητοποίηση, να υπάρχει μια ενσυνειδητότητα δηλαδή. Γιατί αν δεν υπάρχει ζήτηση ελεφαντοστού τότε δεν θα υπάρχει και παρόμοιο έγκλημα, δεν θα προωθεί αυτό το έγκλημα. Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλδημοκράτες. Τον λόγο έχει ο κύριος Πότια. για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους με τους οποίους είχα την ευχαρίστηση να συνεργαστώ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και πραγματικά η προσέλευση στην αίθουσα δεν είναι ανάλογη της σημασίας του θέματος. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ε, όσο άλλοι συνάδελφοι. Πριν από ένα χρόνο στην αίθουσα αυτή συζητούσαμε την, ε, τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπό το φως και εν της διάσκεψης της ε, της συνθήκης ΣΑΙΤΙΣ για τα προστατευόμενα είδη. Γνωρίζαμε όμως πως δεν ήταν μόνο ζήτημα ευζωίας των ζώων, αφορά ολόκληρα οικοσυστήματα και ολόκληρα είδη. Το 2013 είχαμε σοβαρή επιδίνωση της ε, κατάστασης. Εγκληματικές οργανώσεις ε, μπήκαν ε, στο παιχνίδι της εμπορίας τέτοιων παρανόμων ειδών και έφτασε μέχρι να χρηματοδοτείται και η τρομοκρατία από αυτό. Ο ΙΕ έκοψε τον κόνδωνα του κινδύνου, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ζώα και καμιά φορά είναι μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού των ζώων αυτών που αφανίζεται Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν η Κομισιόν σκοπεύει να ρυθμίσει το εμπόριο αυτό στο ίντερνετ. Υπάρχουν πολλά παραθυράκια εκεί. Και επίσης θα ήθελα να ακούσω τι θα κάνει η Κομισιόν για να σταματήσει η εισαγωγή ε, κυνηγητικών τροπέων και άλλων τέτοιων ειδών. Σας ευχαριστώ για τους φιλελεύθερους για 3,5 λεπτά. Τον λόγο έχει ο κύριος Γκέρμπραντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την ε, απάντηση στην ε, ερώτησή μας. Χαίρομαι με αυτά τα οποία μας λέει ο κύριος ε, Επίτροπος, δηλαδή προσεχώς θα έχουμε ανακοίνωση, θα έχουμε διαβούλευση. Ε, δεν φτάνουν αυτά τα πράγματα και κινούνται και πάρα πολύ αργά. 10 Απριλίου η διαβούλευση. Από τώρα μέχρι τις 10 Απριλίου είναι τρεις μήνες. Τρεις μήνες σημαίνει 10.000 ελέφαντες νεκροί. Έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα. Τι ε, μπορούμε να κάνουμε λοιπόν όταν γινόμαστε τόσο αργά. Γινόμαστε τόσο αργά. Καταλαβαίνω αυτά που λέει ο κύριος Ποτότσνικ, αλλά πρέπει πραγματικά να κινηθούμε κάπως διαφορετικά. Είπα εδώ πέρα ε, παίζουν υποδειγματικό ρόλο. Η Χίλαρη Κλίντον ως Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το ζήτημα στην ε, ημερήσια διάταξη σε πανεθνικό εκεί επίπεδο. Ο δε πρόεδρος Ομπάμα στην, επίθεση, στην συγχωρείτε, επίσκεψή του στην Αφρική το ίδιο. Δεν είναι δυνατόν να φερόμαστε έτσι στην ε, άγρια ζωή. Αυτό έχει και τεράστιες κοινωνικέ επιπτώσει στην Αφρική, στην Ασία και σε πολλά μέρη του κόσμου. Και επίσης μην ξεχνάμε πως ε, πλέον μιλάμε για μια τεράστια εγκληματική δραστηριότητα, έτσι. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ε, ζητήσω από τον κύριο Επιτρόπο να κινηθεί ακόμα γρηγορότερα. Όχι μόνο να υπογράψουν ένα μνημόνιο συναντήληψης με τον ε, Κινέζο ομολογό του, αλλά ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το συζητήσει με τον πρόεδρο της Κίνας και με το πρωθυπουργούς ε, στην Αφρική και αλλού. γιατί πρέπει βεβαίως να δούμε τι γίνεται και με τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Μπορούμε όλα αυτά τα παράνομα τα οποία μαζεύονται και κατάσχονται να καούν δημοσίως ε, για να καταστήσει σαφές πως δεν είναι δυνατόν να εισάγονται στις χώρες μας αυτά. Κύριε Πρόεδρε, διάσα χτες πως ο Λέοντας ε, το λιοντάρι εξαφανίστηκε από την Δυτική Αφρική. Ε, στο ίδιο κομμάτι δε πλέον έχουν απομείνει οι τελευταίοι ελέφαντες. Έχουμε πολύ, πολύ λίγο χρόνο. Πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να κινητοποιηθεί. Το 2009 έγιναν συστάσεις στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικό, δεν αφιέρωσαν πόρους, προτεραιότητες στην εξυχνίαση και στην δίωξη αυτού του φαινομένου. Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι πλέον ε, χώρος ε, προορισμού και διακίνησης τέτοιων προϊόντων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Για δύο και μισό λεπτά η κυρία Μπελιέ για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι. Η προφορική αυτή ερώτηση και το ψήφισμα που συζητάμε και θα εγκρίνουμε αυτή την εβδομάδα, ελπίζω με μεγάλη πλειοψηφία, είναι μια έκκληση για την ανταπόκριση σε ένα τεράστιο πολιτικό διεθνές πρόβλημα. Η... Με συγχωρείτε κύριε Μπέλια, μήπως μπορείτε και εσείς πιο αργά γιατί οι διερμηνεύτριες καθυστερούν. Το λαθρεμπόριο φυτών και ζώων είναι το τρίτο μεγαλύτερο μετά από τα όπλα και τα ανθρώπινα όντα. Υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε σχεδόν 30 δισεκατομμύρια το χρόνο. Οι ελέφαντες εξοντώνονται για το ελεφαντοστούν. Στο Καμερούν το 2012 βρέθηκε υπήρχαν λαθροκυνηγοί που προέρχονταν από το Σουδάν σε οργανωμένα, με οργανωμένο τρόπο. Και υπάρχουν και άλλα τέτοια προϊόντα, δόντια τίγρεως, ε, κέρατα ρινοκέρων, τίποτα δεν αφήνουν οι πειρατές της βιοπικιλότητας. Το λαθρεμπόριο αυτό ξεπερνάει τις δυνατότητες και το απλό θέμα της βιοπικιλότητας όμως. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι αυτές οι δραστηριότητες τροφοδοτούν το οργανωμένο έγκλημα διεθνώς την, ε, το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος και ίσως και τρομοκρατικές δραστηριότητες. Έχουν σκοτωθεί και πάρα πολλοί φύλακες αυτή η εγκληματικότητα λοιπόν σιγά σιγά γίνεται μια τεράστια απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια. Η Ιντερπόλ και άλλα διεθνή σώματα έχουν ζητήσει από όλες τις αστυνομίες να καταπολεμήσουν αυτές τις δραστηριότητες και πολλά κράτη προβλέπουν ε, κυρώσεις για τέτοιου είδους δραστηριότητα. Εδώ πρόκειται λοιπόν και για απώλεια της βιοποικιλότητας και για ζημία κατά του περιβάλλοντος αλλά πρέπει κάτι να αλλάξει εδώ γιατί ε, το έδαφος της Ευρώπης είναι το έδαφος από όπου περνούν όλα αυτά τα λαθρεμπόρια και το ψήφισμά μας αυτό στοχεύει ακριβώς να υπάρξουν σοβαρά εργαλεία αντιμετώπισης ζητούμε από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο να δράσουν και να ζητήσουν και συνεργασία με την Ιντερπόλ για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση αυτού του προβλήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία συνάδελφε. Για δύο λεπτά τον λόγο έχει για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς η κυρία Γκέρλινγκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να πω πως ε, εξ ονόματος της ομάδας μου καλωσορίζω το ψήφισμα αυτό. Βεβαίως πρόκειται για μια φρικτή δραστηριότητα και είναι σημαντικό το θέμα και για εμάς. Η λαθροθυρία εμβληματικών ειδών ε, όπως τα λιοντάρια και οι ελέφαντες βεβαίως εξοργίζει τον κόσμο αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα μικρότερα είδη που έχουν μεγάλη σημασία για τη βιοπικιλότητα, που είναι εξίσου σημαντικά. Πρόκειται λοιπόν για ένα περίπλοκο ψήφισμα και δεν έχουμε χρόνο να τα αναπτύξουμε όλα αυτά εδώ. Αλλά ε, η ομάδα μας είναι υπέρ. Τούτου λευθέντος θα ήθελα να φέρω δύο τομείς ε, που ανησυχούν ε, την ομάδα μας. Πρώτον, η έκκληση για εναρμόνιση της νομοθεσίας και η παραγωγή, η δημιουργία κοινών κυρώσεων. Θα ήταν λάθος να δώσουμε τόσο μεγάλη έμφαση στην προσέγγιση αυτή, διότι δεν θα επιτευχθεί εύκολα και μπορεί να οδηγήσει